Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση, Περικέ συμφωνίες με το Μεξικό και τη Χιλή προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικαιροποίηση και τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού και μια δεύτερη προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής. Να δώσω απευθεία το λόγο στον κύριο Μορέιρα, συντάκτη της προφορικής ερώτησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου αυτής, του Κοινοβουλίου, σας παρουσιάζω τις δύο προφορικές ερωτήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή μας. Ε, τις απευθύνουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν το μέλλον των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό και με την Χιλή. Ο Ζορς Κούτας ε, έχει συνυπογράψει την, ε, ε, την ερώτηση για το Μεξικό και η κυρία Ζαμόρα, Θαμόρα που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, δεν τα κατάφερε, συνυπέγραψε την προφορική ερώτηση για τη Χιλή. Ας ξεκινήσω ευχαριστώντας και τους δύο για την αποφασιστική του συνεισφορά για αυτές τις δύο ερωτήσεις και για τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα μετά. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό βασίζονται σε Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, Πολιτικού Συντονισμού και Συνεργασίας που ετέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2000. Ε, σε ό,τι αφορά την Χιλή, ε, οι σχέσεις ε, βασίζονται στη Συμφωνία Σύνδεσης που υπογράφηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002. Πρόκειται για συμφωνίες που χρονολογούνται παραπάνω από 10 χρόνια πριν και όταν υπογράφηκαν ήταν εμπορικές, ε, ήταν από τις πιο προχωρημένες και φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε όμως ε, έχει αλλάξει το ε, πολιτικό περιβάλλον και προς τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ε, πολλές εμπορικές συμφωνίες, διμερείς εμπορικές συμφωνίες και με την Κεντρική Αμερική και με την ε, Κολομβία για παράδειγμα, πρόσφατα με τον Καναδά. Αυτή τη στιγμή ε, διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείες και παραμένουν ανοιχτές διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Το Μεξικό και η Χιλή από την άλλη πλευρά βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την διαειρηνική ειρηνική εταιρική σχέση ε, και μαζί με την Κολομβία και το Περού συμμετέχουν σε ε, διαπραγματεύσεις περιφερειακής ολοκλήρωση ενώ έχουν υπογράψει συμφωνίες και με πολλές άλλες τρίτες χώρες. Σε, αυτή, σε αυτό το πλαίσιο ε, είναι λογικό να σκεφτούμε το πώς μπορούν να εξυγχρονιστούν οι δύο αυτές συμφωνίες. και οι εμπορικοί εταίροι θα πρέπει να το εξετάσουν. Από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εμπορικέ συμφωνίε τελευταία γενιά, ξεκίνησαμε με την Κορέα είναι πολύ πιο φιλόδοξε τόσο σε ό,τι αφορά το πεδίο όσο και σε ό,τι αφορά την, ε, το βάθος της ε, απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. Για παράδειγμα, περιλαμβάνονται οι κρατικέ προμήθειε, δικαιώματα αποτελεσματική διοκτησία, άμεσε εξωτερικέ ε, επενδύσει, Χωρίς να ξεχνάμε το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης ε, με εργασιακές και περιβαλλοντικές ε, ρήτρε, ε, κάτι που πραγματικά πλησιάζει πολύ όλες αυτές τις συμφωνίες στο κοινωνικό κεκτημένο. <clears throat> Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτές οι δύο συμφωνίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εξυγχρονιστούν. Το πρώτο ερώτημα είναι ε, αν θα πρέπει ε, να ενημερωθούν και να διευρυθούν αυτές οι συμφωνίες ή αν θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθούν οι ρήτρες αναθεώρησης, ρήτρα αναθεώρησης της Συμφωνίας του Μεξικού και ρήτρα εξέλιξης συμφωνίας με τη Χιλή. Οι δύο αυτές προφορικές ερωτήσεις έχουν ως στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια αξιολόγηση των εταιρικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ε, Μεξικό για τη Χιλή μετά από αρκετά χρόνια εφαρμογής αυτών των δύο συμφωνιών και επίσης να καταλάβουμε αν το ε, νομικό πλαίσιο των σχέσεων με αυτές τις δύο χώρες χρειάζεται να εξυγχρονιστεί. Ποια είναι τα σημεία κλειδιά μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης ε, και σε πιο χρονικό ορίζοντα. Ε, τέλος, ε, ποια είναι η προτεραιότητα που έχουν αυτές οι δύο χώρες στην διαπραγματευτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Αυτή είναι η βασική στόχη των δύο αυτών ερωτήσεων της ΣΥΝΤΑ και ως ε, μέλος του και ως ε, βουλευτής πλέον ε, εύχομαι η συζήτηση αυτή να πετύχει τους στόχους της. Περιμένουμε να μας απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Κάλλας έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ο Επίτροπος Δεγκούχτ δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εδώ σήμερα για την κοινή συζήτηση για το μέλλον ε, των δύο αυτών μελών της ε, Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου του Μεξικού και της Χιλή. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μου χαρά εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το Μεξικό να ξεκινήσουμε. Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της ΕΠΑ. Και ε, μετά της ΕΠΑ πάλι τρίτος μεγαλύτερος εταίρεο εισαγωγών. Αυξάνονται λοιπόν οι εμπορικέ συναλλαγέ τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατε μεταρρυθμίσει στο Μεξικό δημιούργησαν πολύ ενδιαφέρουσε προοπτικέ για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε σε τομεί όπω οι τηλεπικοινωνίε και άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώ είναι υπέρ τη περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με το Μεξικό και συζητά στην παρούσα φάση με τους Μεξικανούς ομολόγους πώς θα επιτευχθεί αυτό Υπάρχει πλέον συνένεση ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια αναβάθμιση που θα καλύπτει το σύνολο των ε, συμφωνιών με το Μεξικό και να δημιουργηθεί λοιπόν μια κοινή ομάδα εργασίας ε, Ευρώπης και Μεξικού για το σκοπό αυτό. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και τα μέρη αποφάσισαν, ε, έλαβαν αποφάσεις σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, δασμών, γεωγραφικές ενδείξεις, κανόνες ε, για την ε, προέλευση, θέματα φυτοπροστασευτικά, τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Και προβλέπεται μια δεύτερη συνάντηση το Φεβρουάριο στο, στην πόλη του Μεξικό, όπου θα συνεχίσουν να εξετάζουν δυνατότητε εξυγχρονισμού. Βασική τομή σε συζήτηση θα είναι οι δημόσιε συμβάσει, ο ανταγωνισμό, η προστασία των επενδύσεων, το εμπόριο, τα προγράμματα και τα μέσα προστασίας του εμπορίου και η βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. Βάσει λοιπόν των δύο αυτών ε, συναντήσεων θα καταρτιστεί μια κοινή έκθεση η οποία και θα καταγράφει την κατάσταση. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια αξιολόγηση και των επιπτώσεων της ε, σημερινής ε, συμφωνίας και ποιος θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της ενδεχόμενης μελλοντικής σύμβασης και συμφωνίας. Η έρευνα αυτή θα εξετάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και στο Μεξικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά θέματα απασχόλησης, μισθών, εισοδημάτων των νοικοκυρών, μείωση της ένδυας και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επίσης θα αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ιδιαίτερως αυτοί που συμβάλλουν στο πρασίνισμα της οικονομίας. Η μελέτη θα ποσοτικοποιήσει επίσης τα υπόλοιπα εμπορικά προσκόμματα, κυρίως τα βασμολογικα προκειμένου να δούμε πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην εξυγχρονισμένη συμφωνία. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστηθεί, να, να γίνει σύσταση για έναρξη διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από τις διερευνητικές αυτές συνομιλίες με το Μεξικό, από το επίπεδο φιλοδοξίας και από την πληρότητα αυτών, αλλά και από τα αποτελέσματα της εκθέσης ε, αξιολόγησης. Αν αποφασίσουμε να εξυγχρονίσουμε και όταν για να νεώσουμε αυτή τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ενδεχόμενες βελτίωσεις του κεφαλαίου για τις ε, οικονομικές υπηρεσίες και προκειμένου να υπάρχουν σαφείς ε, νομικά δεσμευτικέ δεσμεύσεις. Γιατί χελεί τώρα οι διμερεί ε, εμπορικές ε, διαπραγματεύσει και σχέσεις βασίζονται σε μια πολύ επιτυχή συμφωνία. Από την 1η Φεβρουαρίου του 2003 το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά 128% και έχει φτάσει τα 18,1 δισεκατομμύρια το 2012. Μεταξύ του 2004 και του 2011 οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπηρεσίες στη Χιλή έχουν αυξηθεί κατά 128% ενώ οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 87%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει η βασική πηγή ξένων και αλλοδαπών επενδύσεων. 21,5% στη Χιλή άμεσες επενδύσεις το 2012. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι και, οι δύο, τα δύο μέρη έχουν έντονο οικονομικό συμφέρον να αναπτύξουν περαιτέρω α, τέτοιες διατάξεις και μια ανδεχόμενη ζώνη ελευθερου εμπορίου θα περιλάμβανε διάφορες ε, διατάξεις και διάφορες εμπορικές συμφωνίες που έχουν ε, συμφωνήσει τα μέρη. Για παράδειγμα, Υπάρχει μεγάλη, μεγάλος αριθμός διατάξεων σε ό,τι αφορά ε, την ε, προέλευση, σε ό,τι αφορά φυτοπροσαρτητικά μέτρα, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και αυτά έχουν εφαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο και αυτό ωφελεί και τα δύο μέρη. Η ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση της εμπορικής συμφωνίας η οποία ολοκληρώθηκε το 2012, επαλήθευσε όλα αυτά τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι και το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας θα μπορούσε να ανανεωθεί σε ό,τι αφορά για τις υπηρεσίες, για παράδειγμα, τις ε, επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, τα τεχνικά ε, εμπόδια για τα προστατευτικά μέτρα, βιώσιμη ανάπτυξη και το καθεξής. Και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει ένα non-paper που έχει ως τίτλο «Πρόταση για την ε, εξυγχρονισμό της, ε, σχέσης, της Συμφωνίας Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικό». Και τον Οκτώβριο του 2013 έγινε μια σχετική συνάντηση. Περιλαμβάνονται λοιπόν στο έγγραφο αυτό πολλά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και τα αξιολογεί ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Χιλή σηματοδοτεί ότι είναι πρόθυμη να συζητήσει τους τομείς που δεν καλύπτονται από την αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την γεωργία και τις υπηρεσίες από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα και αυτή να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σαφεί δεσμευτικέ διατάξει και να εξεταστεί βελτίωση του κεφαλαίου για τις οικονομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις νέες ε, την αναμοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τραπεζικό κλάδο. Χρειάζεται λοιπόν έντονη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Είμαστε σε μια προκαταρτική φάση και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Χιλή και θα πρέπει ασφαλώς να συνεχίσουμε τις διαβολεύσεις με τα κράτη-μέλη, με το, με το Ευρωκοινοβούλιο για να εντοπίσουμε τους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για το ΕΛΚ κύριο κύριος για τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να σας πω ότι αυτές οι συμφωνίες δεν είναι συμφωνίες εμπορίου, είναι συμφωνίες σύνδεσης, είναι οι πρώτες συμφωνίες που σύναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν το χαρακτηριστικό ότι ήταν συμφωνίες τέταρτης γενεάς με ε, τρίτες χώρες. Το πρώτο ήταν βιομηχανική συνεργασία, η δεύτερη γενεά ήταν ε, ε, τεχνολογική συνεργασία, η τρίτη ήταν δημοκρατική ρήτρα και η τέταρτη ήταν η ε, σταδιακή βελτίωση των συναλλαγών οι συμφωνίες αυτές ε, είναι ε, η ιστορία μιας επιτυχίας. Ο Επίτροπος μας ε, υπενθύμησε τι θεαματικά αποτελέσματα είχαμε στη συμφωνία με τη Χιλή. Πάνω από 230% κέρδος στη πρώτα χρόνια της εφαρμογής της συμφωνίας με τη Χιλή και πολύ μεγάλη βελτίωση των συναλλαγών και των υπηρεσιών και είχαμε πάνω από 800 δις ευρώ κύκλο εργασιών. Όπως υπενθύμησε ο κύριος Μορέιρα, πριν από μία δεκαετία και όταν ε, ξεκίνησαν αυτές οι συμφωνίες έχουν αλλάξει πλέον οι συνθήκες. Ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τον Καναδά, με την Ιαπωνία, με τη Νέα Ζηλανδία, με την Αυστραλία και με τις ε, χώρες της ευρύτερης γειτονίας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν μεγάλες μελέτες και πάρα πολλές συνεδριάσεις κύριε Επίτροπε για να κατανοήσουμε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν αυτές οι συμφωνίες και πρέπει να επικαιροποιηθούν και να είναι σύμφωνες με τους καιρούς μας. Τον Ιανουάριο πέρσι, πριν από ένα χρόνο κύριε Επίτροπε, συζητήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει εξυγχρονισμό τη συμφωνίε με τη Χιλή. Πέρασε ένα χρόνο, εσεί αναφερθήκατε στην προσφορά τη Χιλή, την οποία παρουσίασε πριν από αρκετού μήνε και εμεί περιμένουμε ακόμα την κατάλληλη απόδειξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση του Μεξικού έχουμε πολύ σημαντικέ συνταγματικέ μεταρρυθμίσει, κυρίω στον τομέα των υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και τη ενέργεια, που θέλουν πραγματικά να ανανεώσουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα υποφεληθούν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα μεγάλο βραβείο γιατί προλαμβάνει τις καταστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι ήγηκε η ώρα να δώσουμε μια απάντηση στην πλευρά της Χιλής και να ε, ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα της εξέλιξης της συμφωνίας και θεωρώ κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση ώστε να υπάρχουν νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ε, βελτίωση της συμφωνίας με το Μεξικό πριν ολοκληρωθεί η θητεία της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτροπής. Ό,τι γίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Επίτροπε, πραγματικά νομίζω ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων των ε, πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε, διότι πέρασε πολύτιμος χρόνος από τότε που ολοκληρώθηκε η διάσκεψη της Χιλής και των δεσμεύσεων που αναλάβαμε και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Κουτάς για ένα λεπτό και τρίαντα δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία Οικονομικής ε, ε εταιρική σχέση πολιτικού συνορισμού και συνεργασία με το Μεξικό έχει προσφέρει ωφελήματα και προς τα, δύο μέρη. Από το, μεταξύ του 1999 και του 2012 οι εξαγωγές ευρωπαϊκών προς το Μεξικό αυξήθηκαν κατά 164% και αντίστροφα ε, κατά 196% από το Μεξικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά διάρκεια αυτής της ε, περίοδου βέβαια ε, οι, οι παγκόσμιες συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχουμε πολλές και πολύ πιο φιλόδοξες τέτοιου τύπου συμφωνίες. Οπότε και οι δύο εταίροι έχουν διάθεση να εξυγχρονίσουν τη συμφωνία αυτή. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, πρόσθετε, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή και να περιλαμβάνει και μια ρήτρα βιώσιμη ανάπτυξη, καθώ επίση ε, και μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει επίση να συμπεριληφθούν και οι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε. Θα ήταν ένα πραγματικά καλό παράδειγμα ε, συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού για την καταπολέμηση της ε, απάτης και της φοροδιαφυγής. Ε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ και έχει υπογράψει συμφωνία με τον Καναδά, θα πρέπει όλε αυτέ οι συμφωνίε να είναι συνεπεί μεταξύ του. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ για του πρασίνου. Δεν είναι πεπισμένη ότι η διεύρυνση ε, με το Μεξικό και την Χίλα είναι ένα, και τη Χιλή σημαντικό βήμα. Ε, ξέρουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Trade ήδη είναι επιβαρημένη με όλες τις ε, διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες ε, που διενεργούνται με χώρες σε όλο τον κόσμο. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Εγώ θέλω να ακολουθήσουμε μια στρατηγική ε, ε, ε, δίκαιου εμπορίου, fair trade. Οι, στατιστικές, οι στατιστικές είναι επίσης ξεπερασμένες, αντιστοιχούν στο 19ο αιώνα. Διαβάστε το άρθρο του Πασκάλ Αμή του Δεκεμβρίου. Λέει ότι οι παγκόσμιες ε, αξίες έχουν αλλάξει. το πάνω από το 60% του εμπορίου είναι στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Ε, μάλλον μεταξύ επιχειρήσεων. Ε, το έχετε σκεφτεί αυτό. Ε, πώς το παγκόσμιο εμπόριο συνάδει με αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Μεξικό. Πόλεμος για τα ναρκωτικά με το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα αυτά τα πράγματα πριν να μαθαίνουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο ε, τη αριστερά, ο κύριο Σόλτ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τι εννοεί το, η ομάδα μου με τον εξυγχρονισμό τη ε, εμπορική συμφωνία. Μεγαλύτερο όφελο για την κοινωνία, κοινά μέτρα για την ενίσχυση των ε, εργασιακών δικαιωμάτων, βελτίωση τη προστασία του περιβάλλοντο και το καθεξής. Όταν ο Επίτροπος μιλά για εξυγχρονισμό, καταλαβαίνει όμως ότι φέτος ε, περαιτέρω φιλελευθεροποίηση. Αν η συμφωνία με τον Καναδά και οι στόχοι διαπραγματευτικοί με τη ΣΥΠΑ αποτελούν το ε, πρόγραμμα και το παράδειγμα για μια τέτοια ε, εξυγχρονισμένη συμφωνία με το Μεξικό, δεν μπορεί να την υποστηρίξει η ομάδα μου αυτή την συμφωνία. Να σκεφτείστε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολε οι συνθήκε που αντιμετωπίζει το Μεξικό και είναι ε, πολύ μεγάλο ο εμφύλιο πόλεμο. Και τα αποτελέσματα τη ναύτα για το Μεξικό θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ βάθρων. Αν δεν προχωρήσετε σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με το Μερκοσούρ, η ομάδα μου δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει μια μεγάλη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Χιλή σε ό,τι αφορά την διαδικασία αυτή ενοποίηση τη Νοτιοαμερική Σήμερα χρειαζόμαστε συμφωνίες συνεργασίας για οικονομική συνεργασία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που θα εξυπηρετήσουν τις κοινωνίες του 21ου αιώνα. Αυτός θα πρέπει λοιπόν να είναι η εντολή για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και από αυτό προκύπτουν οι ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Σινκλέρα πουσιάζει. Επομένως, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Θάλμπα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, η Χιλή και το Μεξικό εδώ και χρόνια αποδεικνύουν ε, την αλληλεγγύη τους ε, και την ε, βιωσιμότητά τους ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των συμφωνιών που έχουν και οι δύο χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάνω περίπου από 20 χρόνια. Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις και με τις δύο χώρες από τότε που συνάφθησαν οι συμφωνίες και είναι σαφές διότι έχουν βελτιωθεί εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Χιλής και Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύει λοιπόν ότι η Ήπειρος αυτή, η Λατινική Αμερική, έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει βέβαια να συνειδητοποιήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια το διεθνέ εμπόριο εξελίχθηκε σε διάφορου τρόπου, όπω για παράδειγμα στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Και εμφανίστηκαν και νέοι τομεί ενδιαφέροντο, όπω για παράδειγμα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ταυτόχρονα η Λατινοαμερικανική Ήπειρος ε, βιώνει μια διαδικασία ολοκλήρωσης όπως ε, φαίνεται και από τη Συμμαχία του Ειρηνικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, τη λεγόμενη συμφωνία TTIP όπως είναι γνωστή η βελτίωση αυτών των συμφωνιών δεν αποτελεί απειλή για τις χώρες αυτές, αντίθετα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να βελτιώσουμε τις συμφωνίες σύνδεσης με τη Χιλή και το Μεξικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι να υποφεληθούμε από τις συνέργειες οι οποίες ε, προκύπτουν από αυτό το νέο γύρο, νέα δημιουργία σχέσεων μεταξύ ε, ημών και της Αμερικανικής Υπήρου. Χρειάζεται βελτίωση και όπως είπε ο καθηγητής Μορέιρα υπάρχει η ρήτρα αναθεώρηση στη συμφωνία με το Μεξικό και η ρήτρα εξέλιξης στην περίπτωση της συμφωνίας με τη Χιλή. Στην ε, περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη κάνει μία μελέτη προκειμένου να δει κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιήσει με ε, τον πιο ιδανικό τρόπο τη ρήτρα αναθεώρησης. Με τη χιλή θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ε, προσαρμόσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις μέσω της αντίστοιχης ρήτρας που υπάρχει στη συμφωνία. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι το εξωτερικό εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει κοινοτήριο μοχλό τη ανάπτυξη, γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σχετικά ζητήματα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κατέφτασε η κυρία Σινκλέρ, επομένως της δω απευθεία το λόγο για ένα λεπτό. Δεν θέλετε να λάβετε το λόγο. Θα μιλήσετε μετά. Εντάξει. Ο κύριος Κορτές. Για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντό τη ε, Λατινική Αμερική η περίπτωση Μεξικού είναι ιδιαίτερη. Ε, είναι ο προτιμόμενο συνομιλητή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Οι επενδύσει και η συνεργασία ε, αποτελεί ατμομηχανή για την οικονομική ανάπτυξη του Μεξικού και τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία Σύνδεσης ε, ε, εταιρική σχέση συγγνώμη, πολιτικού ε, συντονισμού και συνεργασίας αποδεικνύουν το κοινό μας όραμα. Οι οικονομικές συναλλαγές με το Μεξικό συνεχώς αυξάνονται από τις σύννευση συμφωνίες και μετά. Έχουμε μάλιστα εργαστεί από κοινού σε πολλά παγκόσμια ζητήματα, από την ασφάλεια μέχρι την, κατα... μέχρι την κλιματικής αλλαγής, ε, καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, ε, ε, τεχνολογία, έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί είναι οι στόχοι που επετεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μένει πολλής δρόμοι μπροστά μας. Ο εξυγχρονισμός της ε, συμφωνίας αυτής θα αποτελέσει αφορμή για να, ε, να κάνουμε πιο στενές ακόμα τη σχέση μας, αλλά και για να δώσουμε στον εαυτό μας ε, δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης απασχόλησης. Είναι πρωταρχική σημασία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει ε, το μήνυμα ότι ο εξορισμό αυτή τη συμφωνία είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρει ομάδε εργασία που έχουν δημιουργηθεί και θα συναντηθούν στο Μεξικό στι 11 με 13 Φεβρουαρίου να, έχουν, να αποκτήσουν μια διαπραγματευτική εντολή. Αυτέ οι ομάδε εργασία θα πρέπει να ενημερώσουν τόσο και την Μικτή Διακοινωνική Επιτροπή, όσο και την Επιτροπή ΙΝΤΑ, όσο επίση και το Κοινοβούλιο του Μεξικού για, τις, ε, για την πρόοδο και για τον οδικό χάρτη του εξυγχρονισμού. Είναι πολύ σημαντικό το έργο της Διαμεκτής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής και επιμένουν να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική πτυχή. Ευχαριστώ. Grazie, ένα λεπτό. Η συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και της Χιλής ε, ε, έχει ξεπεραστεί από την ιστορία δύο παράγοντες απαιτούν τον εξυγχρονισμό της. Πρώτον, η Συμμαχία του Ειρηνικού ε, από τον Απρίλιο του 2011, Περού, Κολομβία, Χιλή, Μεξικό, για την δημιουργία μιας περιφερειακής οργάνωσης που θα οικοδομει σιγά σιγά μια ζώνη οικονομικής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική με ελεύθερη κυκλοφορία ε, προσώπων, κεφαλαίων, ε, υπηρεσιών και αγαθών. Και ε, δεύτερον, ε, οι, οι καινούριε εμπορικέ συμφωνίε που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλήσατε για, την, για ένα άτυπο έγγραφο για τον εξορισμό της συμφωνίας ή το Μεξικό και η Χιλή έχουν δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία ε, του καινούριου κυβέρνηση στη Χιλή και τη καινούρια Κομισιόν, καινούργιου Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ε, πρέπει να προχωρήσουν σε μια καινούργια εποχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία εξυγχρονισμού των συμφωνιών και η ε, Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Χιλή, ε, τη οποία προεδρεύω, θα σα συμπαρασταθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σινκλέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλή επισκέφτηκα τη χώρα πέρσι και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που έχουμε με τη Χιλή. Συμφωνώ ότι αποδείχθηκε ότι η Χιλή είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και με τις δύο χώρες ε, υπήρξαν ε, ε, μεγάλα ζητήματα στη Χιλή, για παράδειγμα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά έχει πλέον προχωρήσει η διαδικασία εκ του και προσπαθεί να διορθώσει όλα τα, μελλοντικά, τα προηγούμενα λάθη της για το μέλλον. Ένα από τα σημεία τα οποία θα ήθελα να θίξω, διότι συμμετείχα σε μακρέ συζητήσει και όλοι αναφέρθηκαν σε συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Αυτό που αναρωτιούνται είναι τι ακριβώ είναι αυτό που έχουν. αν έφευγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπήρχε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Αυτό ήταν το ερώτημα που μου ετέθηκε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπάρχει απειλή με τους ανθρώπους, ε, ε, για του ανθρώπου με του οποίου εκπροσωπώ. Ε, σκέφτονται ότι αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με διάφορε χώρε. Θα ήθελα κάποιο να μου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ε, Και τώρα να περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου. Οι εμπορικέ σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής είναι εξαιρετικά σημαντικές, ιδιαίτερως λόγω και της οικονομικής ανάπτυξης που επικρατεί στην ε, περιοχή. Και το Μεξικό και η Χιλή είναι αξιόπιστοι εταίροι της ευρωπαϊκή Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και να επεκταθούν οι υφιστάμενες συμφωνίες προς όφελος και των δύο των πλευρών. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι σε ό,τι αφορά τις γεωργικές υπηρεσίες και τις δημόσιες προμήθειες θα είναι σημαντικές ε, οι επιπτώσεις. Πιστεύω ότι οι διμερείς συμφωνίες και διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις. Υπάρχουν πολλοί τομει όπου είναι πολύ καλές οι δυνατότητες εξαγωγής ε, προϊόντων από Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κεντρική και Νότια Αμερική αυτοκίνητα, πετροχημική βιομηχανία και άλλη κλάδη. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον Επίτροπο Κάρλος τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξερευνά διάφορους τρόπους για να εξυγχρονίσει τι εμπορικέ σχέσει με το Μεξικό και τη Χιλή. Δύο χώρε που προωθούν την ελεύθερη αγορά όχι μόνο στη Λατινική Αμερική αλλά και στο πολυμερέ πλαίσιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η διερευνητική ε, διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ φυσιολογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντά μας. Έχουμε διαφορετικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό διαφόρων κεφαλαίων και σε σχέση με την ε, τροποποίηση των συμφωνιών. Προτού λοιπόν ζητήσουμε εντολή για τις διαπραγματεύσεις, θα, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η έκθεση για, τις, ε, για το όραμά μας να είσαστε σίγουροι ότι διεξάγεται μια διαδικασία τεχνικής διαβούλευσης και αυτά έχουν προγραμματιστεί για το 2014. Όταν θα έρθει λοιπόν η στιγμή για πολιτικές αποφάσεις, για τις ε, συμφωνίες αυτές, οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν από την εκάστοτε αρμόδια ομάδα και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή